Καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. Chers collègues, la séance est ouverte. η συνεδρία, αγαπητοί συνάδελφοι. <clears throat> Και είναι η πρώτη μα συνεδρία του 2015. Ω εκ τούτου θα ήθελα να σα απευθύνω τι θερμότερε μου ευχέ σε όλου σα προσωπικά, για εσά, για, για τα αγαπημένα σα πρόσωπα και ευχές για την επιτυχία όλων των εγχειρημάτων στα οποία αποδίεστε, μεταξύ των οποίων και το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, ελευθερίας αλλά και ασφάλειας. Έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο, ο οποίος ξεκίνησε με ένα οδυνηρό τρόπο, γιατί υπήρξε μια επίθεση εναντίον των δημοκρατιών μας, στην καρδιά των δημοκρατιών μας, επλήγει η ελευθερία, επλήγει η ελευθερία έκφρασης. Αυτό θα είναι κάτι που θα δημιουργήσει ένα αίσθημα αντίστοιχο με το ηλεκτροσόκ και οι κυβερνήσει μας θα πρέπει κατεπηγόντως να έχουν μεγαλύτερο συντονισμό και να βρούνε ποια, είναι τα κατάλληλα μέτρα για τα, με τα οποία θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε την απειλή αυτή. Του των λεχθέντων θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα την κυρία Φάμπιαν Jones, η οποία βρίσκεται εδώ δεξιά μου. Η Φάμπια Τζόουνς θα είναι αρμόδια για την γραμματεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Έχει ήδη μια σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία για τα θέματα αυτά και της εύχομαι κάθε επιτυχία. Θα αντικαταστήσει τη Μόνικα Στρασέρ, η οποία έχει αλλάξει καριέρα και τώρα είναι υπεύθυνη του τομέα πρωτοκόλλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην οποία επίσης θέλω ευχηθώ κάθε επιτυχία στον νέο ρόλο της και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την ε, δέσμευσή της και για όλα αυτά τα οποία έπραξε υπέρ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σας φέρω τώρα σε γνώση σας τις αποφάσεις των συντονιστών. Στην συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου καταρχήν διορίσαμε εισηγητές. Η ΓΚΟΕ αναλαμβάνει τη γνωμοδότηση για την έκθεση της Επιτροπής Ίτρε που αφορά τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κύριος Ντονάνο από τους σοσιαλιστές θα αναλάβει μια γνωμοδότηση σε σχέση με μια έκθεση της Επιτροπής ε, Αλίας αλίες και συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης. Ο κ. Φερνάντης επίσης από την ομάδα του ΕΛΚ θα αναλάβει τη γνωμοδότηση επίσης για αλλιευτικά θέματα για την ε, Συμφωνία Εταιρικού Χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κάμπο Βέρντ. Επίσης ο κύριος Ταράντ για τους πράσινους σε μια, θα αναλάβει μια γνωμοδότηση και πάλι της Επιτροπής Αλίας είναι το πρωτόκολλο και συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου. Συμφώνησαν επίσης οι συντονιστές για την ημερομηνία του σεμιναρίου το οποίο θα διοργανώσουμε. 31 Μαρτίου θα λάβει χώρα <clears throat> στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι συντονιστές θεωρούν ότι υπάρχει μια δέσμευση και από τη δική σας πλευρά να είσαστε παρόντες, δηλαδή να μην υπάρχει μια απλώς διακεκομένη παρουσία στο σεμινάριο αυτό. Έχουν αναλάβει τη δέσμευση οι συντονιστές ότι θα μπορούν να είναι παρόντες <clears throat> τα μέλη της Επιτροπής μας από το πρωί ως το απόγευμα, ώστε να είναι και διαδραστικό και καρποφόρο το σεμινάριο αυτό. Θα ήθελα επίσης οι συντονιστές να μου πούνε ποια είναι τα άτομα ή ποιες είναι οι προσωπικότητες καλύτερα που θα μπορούν να προσκληθούν για να μας δώσουν τη μαρτυρία τους και να μας ε, εμπλουτίσουν με τη γνώμη τους σε αυτό το σεμινάριο. Ο κ. Φερνάντες, ο οποίος είναι γενικός συζήτης για το προϋπολογισμό του 2016, για το τομέα 3, μας έχει προτείνει και ένα χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση των κατευθυντηριών γραμμών του προϋπολογισμού του 2016. Ο κύριος Δεπρέ θα είναι ο συζήτης για τα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού. Μας έχει υποβάλει μια ενδιάμεση έκθεση και θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά ως ο νουπο η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα συμμετάσχει επίσης στην Διακοινοβουλευτική Εβδομάδα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου, προβλέπει τη συμμετοχή και τη συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών η Επιτροπή μας θα είναι και αρμόδια για τη διοργάνωση ενός ειδικού εργαστηρίου όπου θα εστιάσουμε τον προβληματισμό μας στα ραλ, στα ποσά τα οποία δεν έχουν εκταμιευτεί, στους λογαριασμούς οι οποίοι παραμένουν εκκρεμείς. Προβλέπεται λοιπόν στη διακοινοβουλευτική αυτή η εβδομάδα να υπάρξουν συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα λάβει χώρα αυτή η συνάντηση στις 3 και 4 Φεβρουαρίου και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε ως το δυνατόν πιο διαθέσιμοι σε αυτές τις ημερομηνίε και να μπορέσετε με τον τρόπο αυτό να αποτελέσετε μια γέφυρα <clears throat> με τους ε, εθνικούς κοινοβουλευτικούς που θα είναι παρόντες εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη συντονιστική διαδικασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Εγώ ίδιος έχω συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία ως εθνικός κοινοβουλευτικός σε αυτές τις εβδομάδες και πρέπει να σας ε, ομολογήσω ότι έχω νιώσει μια μεγάλη ματέωση στο παρελθόν σε σχέση με τον, και με τον τρόπο τον όχι ιδιαίτερα οργανωμένο τρόπο συζήτησης που, οδήγησε, που δεν οδήγησε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και εμείς από τα Εθνικά Κοινοβούλια είχαμε πολλές δυσκολίες για να εξηγήσουμε στους ομολόγους μας <clears throat> το πώς είχαν λειτουργήσει αυτές οι εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Τώρα, οι αποφάσει που ελήφθησαν σήμερα το πρωί, γιατί πριν από τη συνεδρίαση τη Επιτροπή μας έλαβε χώρα μια συνεδρίαση των συντονιστών, αποφασίσαμε να συντάξουμε μια γνωμοδότηση για μια έκθεση πρωτοβουλία τη επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων, Συνταγματικών Θεμάτων, σε σχέση με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την συνθήκη της Λισαβόνας. Και ο πρόεδρος σας ο ίδιος, η ταπεινότητά μου, έχει διοριστεί ως εισηγητής για την γνωμοδότηση αυτή. <clears throat> Αποφασίσαμε επίση να έχουμε μια γνωμοδότηση για μια έκθεση πρωτοβουλία τη Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων, Ρέτζι, Πρόκειται για τις επενδύσεις για την ε, απασχόληση και την ανάπτυξη. Η πρόθεση της οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σοσιαλιστική ομάδα η οποία θα αναλάβει αυτή τη γνωμοδότηση. Για την γνωμοδότηση αυτή λοιπόν και για την έκθεση της Επιτροπής ΙΝΤΑ, μακροδημοσιονομική αρρωγή προς την ε, Ουκρανία, <clears throat> θα εκδώσουμε γνωμοδότηση, ούτε για την έκθεση της ΛΥΜΠΕ, για την ενδιάμεση έκθεση και τον Ευρω... για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Για το σχέδιο τώρα επενδύσεων της Κομισιόν. Το σχέδιο δηλαδή που κατέθεσε ο κύριος ε, Γιούγκερ, οι συντονιστές μας όταν συσκέφθηκαν αποφάσισαν να διατηρήσουμε τον ηγετικό ρόλο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για τη νομική βάση. Οι υπόλοιπε επιτροπές είναι συνδεδεμένες επί τη βάση του άρθρου 54 του κανονισμού ΕΚΟΝ, ΤΡΑΝ, ΙΤΡΕ και κατά πόσα πιθανότητα και άλλες επιτροπές θα είναι συνδεδεμένες. Προσπαθήσαμε να αντλήσουμε διδάγματα από την διαδικασία ε, έγκρισης ε, του προϋπολογισμού για το δεύτερο εξάμεινο του 2014 και επίση να συνειδητοποιήσουμε γιατί ήταν τόσο απογοητευτικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής της συνθήκη της Λισαβόνας για τα δημοσιονομικά ζητήματα. Συντάξαμε ένα έγγραφο το οποίο κατά τη γνώμη μας θα λειτουργήσει ως βάση για το σεμινάριο του Μαρτίου, ε, θα γίνει το Μάρτιο στις 31. Για την Επιτροπή μας οι συντονιστές αποφάσισαν τις ημερομηνίε για τα ταξίδια, τις αποστολές. Ουκρανία, ε, εβδομάδα 12, 16 έως 20 Μαρτίου. Αυτή η αποστολή θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Εσθονία, εβδομάδα 25. 18 και 19 Ιουνίου. Δύο μέρες μόνο. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για αυτή την αποστολή. Ιταλία, Λαπεντούσα, εβδομάδα 30, 20 με 24 Ιουλίου, τρεις ημέρες θα διαρκέσει θα, ε, ε και η ώρα με τα, του ταξιδιού συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις τρεις ημέρες. Για το Blending and External Cooperation κρίνουν οι συντονιστές ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις των εξωτερικών οργανισμών που συμβάλλουν στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ως προς τα νέα χρηματοδοτικά μέσα Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει το σχέδιό της. Για τις πράξεις εξουσιοδότηση που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν οι συντονιστές μας ότι οι μόνιμοι εισηγητές και άλλοι εισηγητές έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν τις πράξεις εξουσιοδότηση και ότι δεν χρειάζεται να διοριστεί ειδικό εισηγητή για τι πράξει κατεξουσιοδότηση. Ιδού. Αυτέ ήταν οι αποφάσει των συντονιστών. Θα ήθελα. Επίσης να σας ενημερώσω για την κοινοβουλευτική εβδομάδα, α, το έκανα αυτό, 3 και 4 Φεβρουαρίου, κυρίως στις 3 Φεβρουαρίου, μην ξεχνάτε θα γίνει στριγκλή τράπεζα, ε, όπου συντονιστικό ρόλο θα έχει η Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Και φυσικά θα έρθουν όλοι οι βουλευτέ ε, που ασχολούνται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, ε, και ας με διορθώσει η κυρία Γκρέσλε, αν κάνω λάθο, οργανώνουν μία ακρόαση για την απαλλαγή 2013. Την πέμπτη το πρωί θα γίνει αυτό. Έτσι δεν είναι. Η Επίτροπος ε, Γεωργίβα θα παραστεί θα εκπροσωπηθεί και το ελεγκτικό Πέμπτη πρωί, 9 η ώρα στην 5G3 του ΑΣΠ. Πρόεδρε, ε, νομίζω ότι ε, είμαστε και εμείς ευπρόσδεκτοι, έτσι δεν είναι, σε αυτή τη συνεδρία. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω να έχω άλλες ανακοινώσεις. Για τα πρακτικά, για τις συνεδρίες στις 11 και 15 Δεκεμβρίου δεν νομίζω να υπάρχουν ενστάσεις, άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά. Πολύ ωραία. Προϋπολογισμός 2016. Στην ώρα μας αρχίζουμε τη συζήτηση για το τμήμα 3 συγκεκριμένα. Θα δώσω το λόγο στο γενικό μας εισηγητή, τον κύριο Φερνάντες. για να μας παρουσιάσει το όραμά του που θα πλαισιώσει την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2016. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το 2016 θα χρειαστούμε την αφοσίωση και την προσήλωση ολονών, όλων των πολιτικών ομάδων. Αυτό επιθυμώ. Επίσης θα πρέπει να επιδιώξουμε να μετάσχουν ενεργά οι πολίτες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι σημαντικό να αντιληφθούν τη σημασία της διαδικασίας κατάρτισης και υλοποίηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται σε ένα ποσοστό του ΑΕΠ αλλά που προσθέτει, προσφέρει μάλλον μια πάρα πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία. Αυτό πρέπει να επιδιώξουμε. Η, να υπάρξει μια καλύτερη αντίληψη της σημασίας του προϋπολογισμού και να περάσει αυτό το μήνυμα στους ψηφοφόρους, στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 2016, πειθαρχία, αξιοπιστία, είναι, εξακολουθούν να είναι τα σλόγγαν μας. Για τις συμβαστικές λύσεις ε, που θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, Θα πρέπει να είμαστε σαφείς και κυρίως να ε, τη στηρίζουμε κατά την εφαρμογή. Στα πλαίσια τώρα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαίσιου έχουμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και χρειάζεται μία διεξοδική περιστατωμένη εξέταση αυτών των στόχων για να έχουμε την αξιοπιστία. Να χρησιμοποιήσουμε επίσης την προστάμενη αξία του προϋπολογισμού για την υλοποίηση των στόχων αυτής της πολιτικής Ευρώπη 2020 που ενέκρινε η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Για τις προτεραιότητές μας, το μήνυμά μας θα πρέπει να είναι απλό για να γίνει αντιληπτό από τους πολίτες. Τα τρία S στα πορτογαλικά τουλάχιστον, τώρα στη μετάφραση θα έχουμε πρόβλημα. Πρόκειται για την απασχόληση, για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα. Λοιπόν, αυτές οι τρεις έννοιες συνεπάγονται ότι προωθείται και η παιδεία, η επαγγελματική κατάρτιση, η αποσπήρωση της ε, στήριξης ε, που επιφυλάσσεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Α, βγήκε στα γαλλικά η μετάφραση με τα 3 S ε, με το ίδιο γράμμα. Τα τρία ε. Λοιπόν, ε, λοιπόν, και η καινοτομία. Πέραν από αυτό ε, θα χρειαστούμε καλύτερες δεξιότητες, καλύτερη στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, το, η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος επίσης χρειάζεται για δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του προγράμματος μας θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα πιλωτικά προγράμματα με προτεραιότητα την απασχόληση. Έχουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες και δικαίω για τη νεολαία. Επίσης, κινητικότητα αυτών που είναι πάνω από τα 30, έχουμε εκατομμύρια κενές θέσεις απασχόλησης και παραδόξως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνουμε να τις καλύψουμε. Πιστεύω λοιπόν πως αυτό είναι το βασικό μας μήνυμα. Υπάρχουν όμως άλλα δύο. Αυτό της εσωτερικής και της εξωτερικής αλληλεγγύης. Εσωτερική αλληλεγγύη τι σημαίνει. Κοινωνική συνοχή, εδαφική συνοχή και η εξωτερική αλληλεγγύη που σημαίνει καταπολέμηση της ένδυας. Η εσωτερική αλληλεγγύη εξωτερική συγγνώμη, αλληλεγγύη, πολιτική της γειτονίας μας βοηθούν να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο. Έτσι θα αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την κατάσταση στην οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε λοιπόν αναφερθεί πλέον συνοπτικά σε όλες τις προτεραιότητες, αλλά να μην ξεχνάμε ότι Χρειαζόμαστε μια ασφαλή Ευρώπη ταυτόχρονα. Η καλύτερη ε, οικονομία του κόσμου, η ευρωπαϊκή, ε, με... Ε, ε, που υποστηρίζει αξίες όπως ε, η ανεξιθρησκεία, ο σεβασμός, ε, η ανεκτικότητα. Έχουμε το 7% του παγκοσμίου πληθυσμού, όμως δεν έχουμε αντίστοιχα. Έχουμε πολύ ψηλές κοινωνικές δαπάνες σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Θα πρέπει να μην χάσουμε τον προσανατολισμό, τον βασικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το χρονοδιάγραμμα. Στις 5 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών θα παρουσιαστεί το σχέδιο, 11 Φεβρουαρίου για τις τροπολογίες. Στην Επιτροπή θα γίνει ψηφοφορία στις 26 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια θα περάσει το Μάρτιο η έκθεση. Αυτές είναι οι προτάσεις μου, όπως καταλαβαίνετε. Όμως όπως είπα στην αρχή της παρέμβασής μου, βασίζομαι στην συμμετοχή όλων των πολιτικών ομάδων, βασίζομαι στη συμβολή τους, θέλω να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες όλων. Ε, δεν πρέπει όμως να χάσουμε τα ουσιαστικότερα στοιχεία θα πρέπει δηλαδή να εστιάσουμε την προσοχή μας σε, κάποια, σε κάποιες έννοιες κλειδί που εξυπηρετούν το γενικότερο προσανατολισμό που έχουμε υιοθετήσει για τον προϋπολογισμό 2016. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγήτα για αυτή την παρουσίαση που μας κάνατε για αυτά τα... Για τα στοιχεία τα οποία ε, χαρακτηρίζουν τον προπολογισμό για το 2016 και τώρα θα ξεκινήσουμε με μια τελεγή απόψεων για αυτούς τους γενικούς προσανατολισμούς. να λάβουμε υπόψη μας και το σχέδιο Juncker σε αυτό τον προπολογισμό του 2016 που υποτίθεται ότι θα δώσει όθηση στην απασχόληση, ε, στην ανάπτυξη ε, και στις επενδύσεις. Ποιος θέλει να λάβει πρώτο το λόγο? <clears throat> Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ. Εγώ με ο σκιώδης εισηγητής για την σοσιαλιστική ομάδα. Καταρχήν, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φερνάντης για όλα αυτά τα σημεία τα οποία ανέφερε. Είναι οι προτάσει του προτάσει οποίε μπορούμε να συμμεριστούμε, θεωρούμε ότι είναι λογικέ και απαραίτητε. Βέβαια, η απόχρωση που δίνουμε και ο η έμφαση που θα δώσουμε ίσως είναι διαφορετική από τη δική μας πλευρά. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει το θέμα αυτό των κινήτων για μεγαλύτερη κινητικότητα. Αλλά το ερώτημα είναι τι μορφή πρέπει να πάρουν αυτά τα κίνητρα. Εμείς ως σοσιαδημοκράτες θεωρούμε ότι η κινητικότητα πρέπει να σημαίνει ότι ο καθένας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίνει η εσωτερική αγορά και αν έχει το ενδιαφέρον ή αν έχει τη θέληση να δοκιμάσει τις ικανότητες του κάπου αλλού, να το πράξει, αλλά υπάρχει και η άλλη εκδοχή, αν κανείς το κάνει μονάχα αναγκαστικά, επειδή τον υποχρεώνει οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα του. Αν είναι κάτι το οποίο προκύπτει από κοινωνική κατάσταση ανάγκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει μια ελεύθερη επιλογή σε αυτή την περίπτωση. Αυτό δεν μπορεί να είναι λοιπόν η λύση για τα προβλήματα απασχόλησης παρά μόνο σε ένα πολύ περιορισμένο βαθμό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ανισομέρειες στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ορισμένα κράτη <clears throat> τα οποία έχουν ανάγκη για εργασόμενους, έχουν κενές θέσεις εργασίας, αλλά έχουν μεγάλη ανεργία. Η λύση όμως για την ενεργεία για τις τελευταίες χώρες δεν είναι η υποχρεωτική αυτή κινητικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει από άτομα που δεν έχουν άλλη επιλογή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να τους υποχρεώνουμε γιατί δεν θέλουμε να προβούμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι μέσα στον προϋπολογισμό εμείς θα πρέπει να έχουμε την σωστή ε, έμφαση που θα δώσουμε. Αυτό δεν θα αλλάξει βέβαια τα οικονομικά στοιχεία, αλλά πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε απασχόληση μεταξύ των νέων, να δημιουργήσουμε ένα, πλέο, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν οι νέοι και όλοι οι άλλοι να χρησιμοποιήσουν τις ε, δεξιότητές τους. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας εκπλήξει. <clears throat> Είναι και οι προτάσεις οι οποίες είχαμε ήδη διατυπώσει εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει καταρχήν εμείς να υπερασπιστούμε όλες αυτές τις προτεραιότητες που έχουμε διατυπώσει έναντι του Συμβουλίου και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την ευκαιρία της κοινοβουλευτικής εβδομάδος να υπενθυμίσουμε και στα, στους συναδέλφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια την ανάγκη το Συμβούλιο να δώσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τον τομέα της έρευνας, για τον τομέα της ανάπτυξης <clears throat> και της απασχόλησης, γιατί το Συμβούλιο πολλές φορές αναφέρει τα θέματα αυτά, αλλά μετά όταν έρχεται στη διαδικασία του προπολογισμού περικόπτει τα κονδύλια. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο και να καταδείξουμε τις αντιφάσεις στη στάση που παρουσιάζει εναντί του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κολμέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά που είπε ο κύριος Φενάντες είναι έγκυρα και σωστά. Και εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα σαφές ποια είναι η δική μας αντιμετώπιση και η προβληματική μας για τα θέματα αυτά. Έχουμε ακούσει πολλά για πολιτικούς στόχους, έχουμε ακούσει πολλά και για τις τεχνικές πτυχές των θεμάτων αυτών και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε μια μεγάλη συνένεση πέρα από τις πολιτικές παρατάξεις. Λέμε όλοι ότι θέλουμε να αναλάβουμε μέτρα για τη μείωση της ανεργίας των νέων, θέλουμε να έχουμε καλύτερη κατάρτιση, όλα αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Αλλά εδώ πιστεύω ότι το έργο μας θα πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του προϋπολογισμού για το πώς θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν αυτές οι ενέργειες. Γιατί όποιοι στόχοι τίθενται θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν κάποια στιγμή. Αλλιώς είναι απλώς χήμερες τις οποίες εμείς δημιουργούμε, αλλά οι οποίες δεν θα αλλάξουν τίποτα. Δεν πρέπει να έχουμε εγχειρήματα τα οποία δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε στα συγκεκριμένα, στα ψηλά του προπολογισμού, να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα προπολογισμό ο οποίο είναι εξισορροπημένο. Όλοι, όλοι λένε ότι είναι ισοσκελισμένο ο προπολογισμό, αλλά αυτό βλέπουμε ότι είναι μονάχα στα χαρτιά. Γιατί όποιο κοιτάξει καλύτερα βλέπει ότι υπάρχουν χένουσε τρύπε στον προπολογισμό. Το πρόβλημα αυτό τώρα λοιπόν των ποσών που δεν έχουν εκταμιευθεί, των λογαριασμών που δεν έχουν πληρωθεί, αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Και αυτό συνδέεται με το ύψος του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την ίδια άποψη για το θέμα αυτό και το είδαμε στη διαδικασία του προϋπολογισμού, συγγνώμη. Πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Το προπολογισμό που εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο προτάσει της Κομισιόν θα πρέπει να είναι επαρκής για τους στόχους μας. Θα πρέπει λοιπόν το 2016 να εξασφαλίσουμε για τον προϋπολογισμό του 2016 μια έγκαιρη συνεννόηση με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αίσια διαδικασία για τον προϋπολογισμό. Πολλές φορές λένε για μας, για το κόμμα μας, ότι είμαστε επικριτικοί έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι καθόλου κακό για την Ένωση την Ευρωπαϊκή να υπάρξει μια συμφωνία, ε, μια πρώιμη συμφωνία με τα κράτη-μέλη για την οποία θα μπορέσουμε την οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε για τις διαπραγματεύσεις, γιατί σίγουρα αυτό θα οδηγήσει σε μια καλύτερη Ευρώπη. Ο κύριος ε, Μασκά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε ο εισήτης ο κ. Φερνάντζης και οι άλλοι συνάδελφοι εγώ πιστεύω ότι ο κύριος στόχος μας, η κύριη μας προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε όλους τους στρατηγικούς στόχους που θέτουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Γι' αυτό όλε οι ενέργειέ μα θα κινηθούν προ την κατεύθυνση αυτή. Θυμόμαστε όλοι τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν με την ε, χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων μας όταν τα εθνικά κράτη δεν είχαν στον προϋπολογισμό τους απαραίτητους πόρους για συγχρηματοδότηση. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών επί τη βάση μιας εταιρικής σχέσης που θα εξυπηρετήσει το στόχο της Ευρώπης 2020. Αυτό θα είναι μια ευφυής συγκέντρωση των πόρων μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να αντιμετωπίσουμε και τα ελλείμματα των εθνικών προϋπολογισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τους γενικούς ανατολισμούς του Γενικού Εισηγητή. Νομίζω ότι σε αυτά τουλάχιστον δεν ε, υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση. Όμως το θέμα που τίθεται είναι τον, ε, τα μέσα τα οποία πρέπει να διαθέτουμε προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους στόχους. Και εγώ πραγματικά δεν μπορώ να δω πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στους στόχους αυτούς με τα κονδύλια που έχουμε σήμερα. Θα πρέπει να γίνουν ε, κάποιες αλλαγές και θα πρέπει κάπως ε, να τις ε, υποστηρίξουμε αυτές τις μετατροπές. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα σήμερα. Και επομένως το ερώτημα που τίθεται είναι το θέμα των πόρων. Με ποιους πόρους θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε αυτούς τους στόχους με τους οποίους εν γέννη συμφωνούμε θα μπορούσαμε ίσως ε, να έχουμε νέους πόρους, θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε μια κάποια μεγαλύτερη ευελιξία. Πρόκειται για ερωτήματα τα οποία σίγουρα πρέπει να τεθούν και ε, θεωρώ ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στο θέμα των πόρων, στο θέμα της συμμετοχής των κρατών μελών, στο θέμα των νέων πόρων και της ευελιξίας. Και θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση ε, και στην ουσία για τη χρηματοδότηση των Γενικών Προσανατολισμών. Θα είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα και θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια μάχη. Η κυρία Τυρίαντα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την άποψη των υπολείπων και θεωρώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα όπως ε, χωρών όπως η Ιρλανδία που πλήρωσε το τίμημα της λιτότητας και ακόμα πληρώνουμε και είναι πολύ μεγάλο το τίμημα και για κάθε άντρα, γυναίκα και παιδί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν άλλες περικοπές ε, στη συνέχεια, κυρίως για την Αλία που είναι ε, αυτή τη στιγμή κατεστραμμένη στην Ιρλανδία, κυρίως στις μικρές λευτικές κοινότητες και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προσδώσουμε περισσότερη ουσία στη συζήτηση και θα ήθελα να δω πώς ε, θα επηρεάσει το σχέδιο Juncker τον προπολογισμό του 2016 λίγο πιο αναλυτικά, διότι δεν μπορούμε να τα δούμε ξεχωριστά αυτά, είναι αλληλένδετα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τριάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα ακούστηκαν από τον εισηγητή και με τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Ένα από τα σημαντικά κατά την άποψή μου είναι να καταλήξουμε σε συνένεση και να μην ε, ε, φτάσουμε σε αυτό που είχαμε πέρσι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προκειμένου να γίνει δεκτό το σχέδιο προπολογισμού να ξεκινήσουμε νωρίτερα τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη και με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, εάν μου επιτρέπετε. Και επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και το σχέδιο επενδύσεων του Γιούγκερ, διότι θεωρώ ότι η αρχή του επενδυτικού σχεδίου θα είναι εντός του 2016. Επομένως, θα πρέπει να ε, υπάρξουν όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις και συνεργασία ε, στην συζήτηση για τον προπολογισμό του 2016. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάρον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως. Ο κύριος Φερνάντες μας παρουσίασε καλά τη ραχοκοκαλιά των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν για τον προπολογισμό του 2016 και νομίζω ότι θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Το 2015 θα γίνει μια διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να λάβει αποφάσεις που μπορεί και ελπίζω να έχει και θετικές συνέπειες για τον προπολογισμό μας το 2016. Και ίσως θα έπρεπε κατά την κατάρτιση του προπολογισμού για το 2016 να εξετάσουμε και την κατάσταση για την ε, Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση δεδομένου ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι σε ενδιαφέροντα επίπεδα και από τις ενδείξεις που έχουμε από τη ρωσική κυβέρνηση για την ε, ε, κατεύθυνση, ανακατεύθυνση του φυσικού αερίου ή οτιδήποτε σκοπεύουν να κάνουμε το φυσικό αέριο. Όλα αυτά θα έχουν συνέπειε για το μελλοντικό προπολογισμό και θα μπορούσαμε να τα εξετάσουμε και νομίζω ότι έτσι θα καταλάβουν και οι πολίτες τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο Γενικός Εισηγητής θα μας κρατά ενήμερος λοιπόν για τη συνέχεια. Όντως η συζήτηση για τον προπολογισμό που έγινε μετά τις εκλογές ε, του Μαΐου ε, ήταν αρκετά περιορισμένη, ε, χρειάστηκε πολύ γρήγορα να περάσουμε στο τελικό στάδιο και δεν φάνηκε πουθενά και στις συζητήσεις μας αλλά και στο πώς αυτά ερμηνεύτηκαν στη συνέχεια στον προπολογισμό ε, τι ακριβώς δεσμεύσεις αναλέβαμε λόγω της προεκλογικής εκστρατείας. Η μετανάστευση, επί παραδείγματι, ήταν ε, ένα από τα κέρια ζητήματα και ε, η, τα μέσα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι πολύ λίγα. για το Frontex τι έχουμε, ένα εκατομμύριο και αφήνουμε την Ιταλία και την Ελλάδα 80 εκατομμύρια. Την Ιταλία και την Ελλάδα να προσπαθούν να βρουν λύση μόνοι τους. Ή για παράδειγμα το θέμα των νέων. Ε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ορισμένε φορέ έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ανακοινώνουν μεν μέτρα, αλλά δεν εγγράφουν κονδύλια στον προπολογισμό για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα. Και όσον αφορά ε, το θέμα τη εγγύησης για την νεολαία και τους νέους θα ίσως έπρεπε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και να διευκολύνουμε για παράδειγμα την κινητικότητα νέων που κάνουν μαθητεία ε, ή νέων που να μπορούν να μετακινηθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να κάνουμε τέτοιες προτάσεις λοιπόν στο Γενικό Εισηγητή. Όσον αφορά το θέμα των πληρωμών, θα επιμένω στην ε, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, στη Διακυβουλευτική ομάδα. Θα έχουμε εκπροσώπους από διάφορες ε, ε, χώρες, εκπροσώπους των κοινοβουλίων των διαφόρων χωρών και ίσως είναι μια ευκαιρία να τους πούμε ότι όταν συζητούμε τα εθνικά οικονομικά δεν θα πρέπει να μείνουν υπόλοιπα προς εκαθάριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να φροντίζουν να προωθούνται τα κονδύλια. Έχετε κάτι άλλο να πείτε κύριε Σιγητά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, ε, για τη συμβολή τους. Νομίζω συμφωνούν με το πλαίσιο το οποίο έθεσα για τις διαπραγματεύσεις. Πάντως για να τονωθεί η απασχόληση θα πρέπει να ενισχυθεί και η εσωτερική αγορά και η κινητικότητα και κατά την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών μπορούμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πιο κατάλληλα προσαρμοσμένες θέσεις εργασίας, επίσης να κατευθυνθούμε προς την ενεργειακή αυτονομία κατά την αντιμετώπιση του προβλήματος ανεργίας. Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι χρειάζεται συμπληρωματικότητα ανάμεσα στους εθνικούς προϋπολογισμούς αφενός και τον ευρωπαϊκό αφετέρου και Φυσικά συμφωνώ για την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών. Θα ήθελα να πω ε, κάτι για το σχέδιο Juncker. Θελημένα δεν αναφέρθηκα σε αυτό στην αρχική μου παρέμβαση. Σε καμία περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό το επενδυτικό σχέδιο ως ε, κάτι που αντικαθιστά τον ε, προϋπολογισμό. Ε, δηλαδή θα κόβουμε από τον προϋπολογισμό από κάποια κατηγορία, ούτως ώστε λιθαράκι λιθαράκι να αυξάνεται η χρηματοδότηση που έχουμε στο επενδυτικό σχέδιο Juncker. Όχι σε καμία περίπτωση είναι κάτι συμπληρωματικό και θα πρέπει να εξυπηρετήσει το στόχο που έχουμε και εμείς θέσει. Σε καμία περίπτωση όμως και το τονίζω δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ξεκάθαρο πω τα μέσα που χρειαζόμαστε, τα μέσα που χρειαζόμαστε για να υλοποιηθούν οι στόχοι μας θα πρέπει να εξευρεθούν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Όταν όμως μιλάμε για την σαφήνεια, την αξιοπιστία και την τήρηση των δεσμεύσεών μας, ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι χρειάζονται κάποιοι πόροι που θα πρέπει να είναι σε, στη διάθεσή μας. Εάν τώρα δημιουργηθεί κάποια αντίφαση, σίγουρα δεν θα ευθύνεται το Κοινοβούλιο, θα ευθύνεται κάποιο άλλο θεσμικό όργανα. Δηλαδή, θέλω να πω πως ε, έχουμε κάποιες φιλοδοξίες, θέλουμε να υλοποιήσουμε κάποιους στόχους και σίγουρα στις δικές μας τις προτάσεις ε, θα εισηγηθούμε να υπάρχουν τα απαιτούμενα μέσα για την ε, εκπλήρωση αυτών των στόχων. Αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους. Στο σχέδιο που θα καταθέσω δεν θα είναι μυθιστόρημα, έτσι σας καθησυχάζω, θα είναι πάρα πολύ απλή η διατύπωση και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω τα απαιτούμενα στοιχεία με τρόπο όμως που θα γίνει αντιληπτός από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, είμαστε αδίμονες να σας ξαναβρούμε στις αρχές Φεβρουαρίου για να δούμε και το σχέδιο έκθεσή ε, σας. Περνάμε τώρα στα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού, ο εισηγητής είναι ο είναι απόν σήμερα, αλλά εκπροσωπείται από Ιραλή. Δεν προβλέπει ο κύριος Δεπρέ να παρουσιάσει κάποια, κάποιο κείμενο έκθεσης όπως αυτό του κυρίου Φερνάντες, αλλά θα παρουσιάσει παρόλα αυτά ένα έγγραφο εργασίας το οποίο θα περιέχει εκτιμήσεις, προβλέψεις, πρώτες αξιολογήσεις. Θα πρέπει να συναντηθεί και με το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα των άλλων τμήματων του προπολογισμού. Ενδεχομένω ο κύριο Σαλή έχει να μα δώσει συμπληρωματικέ πληροφορίε για τα θέματα αυτά. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, η παρουσίαση του σχεδίου εγγράφου εργασία θα γίνει το Φεβρουάριο στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών μας και η τελική μορφή θα πρέπει να είναι έτοιμη στις 26 Φεβρουαρίου Θα ήθελα να ζητήσω βέβαια εξ ονόματο του κ. Ντεπρέ από τις πολιτικές ομάδες να ε, υποδείξουν ποιοι θα είναι οι σκιώδεις εισηγητές του για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Μασκά, Μανκά. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια ορθολογική λειτουργία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι το οποίο είναι κατεπήγον από την οπτική γωνία της κοινοβουλίας είναι να εξασφαλίσουμε πάντα την ε, έγκαιρη μετάφραση των εγγράφων. Γιατί δημιουργείται πρόβλημα όταν δεν υπάρχει έγκαιρη παρουσία μεταφράσεων. Και επίσης ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία γιατί πολλές φορές μεταφράζεται ασκόπως σε όλες τις γλώσσες ένα έγγραφο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει ότι τα έγγραφα μεταφράζονται μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Ώστε να εξασφαλίσουμε ότι από τη μια μεριά θα έχουμε εγκαίρως τα έγγραφα στη δική μας ε, γλώσσα και να μην καθυστερούν οι μεταφράσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να μην μεταφράζονται άσκοπα έγγραφα και με τον τρόπο αυτό να καθυστερεί η μετάφραση των άλλων. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Δελανό. Ναι, προφανώς. Αν δεν έχουμε τα έγγραφα στη μητρική μας γλώσσα, δεν μπορούμε να υποχρεωθούμε να ψηφίσουμε μια έκθεση. Εγώ σας προειδοποιώ για το θέμα αυτό, το οποίο είναι ένα θέμα αρχής, ένα θέμα ουσίες. Όλοι προσπαθούμε να μιλάμε κάπως αγγλικά και να συνεννοούμαστε, αλλά πρέπει να έχουμε πραγματικά για τα θέματα τα οποία είναι ιδίω σημαντικά τη μετάφραση στις εθνικές μας γλώσσες. Βεβαίως, το ξαναλέω, θα ληφθεί υπόψη αυτό το οποίο ζητήσατε. Ο κύριος Ιτουγάρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο σχόλιο σε αυτό που έλεγε ο συνάδελφος, τον οποίο βεβαίως ε, κατανοώ και συμφωνώ και εγώ μαζί του. Θα ήθελα όμως να κάνω την εξής ερώτηση. Ποιος αποφασίζει ε, ποιο είναι το σημαντικό και ποιο δεν είναι το σημαντικό σε ένα έγγραφο. Γιατί για σας μπορεί να είναι κάτι σημαντικό και για μένα να μην είναι ή το αντίστροφο. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, λίγο περίπλοκης κατάστασης. Ποιος θα κάνει το διαιτητή εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να μου απαντήσει και σε αυτό ο συνάδελφος. Κύριε Μάνκα, θέλετε να απαντήσετε. Ε, ε, είναι σημαντικά αυτά. Ναι, ναι, συμφωνώ με αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν πάντα τέτοια προβλήματα. Εμφανίζονται 700 τροπολογίες σε ορισμένε περιπτώσεις, από τις οποίες 600 τροπολογίες δεν ευδοκιμούν και επομένως δεν μας ενδιαφέρουν και μια εβδομάδα μετά εμφανίζονται μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες. Γι' αυτό <clears throat> θέλω να τονίσω, πρέπει να μεταφράζονται μόνο τα έγγραφα τα οποία είναι ουσιαστικά. Και πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ε, φροντίστε να γράφετε και να λέτε σημαντικά μόνο. Εγώ λοιπόν πρέπει να συγκρατούμε. Ωραία, θα τα υποβάλουμε όλα αυτά στον κύριο Ντεπρέ και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο σημείο υπαριθμών 8. Είναι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αρμοδιότητας της κυρίας Γκορδιαθαμπάλ. Ε, αυτό θα το συζητήσουμε το απόγευμα με την ε, παρουσία της κυρίας ε, Γεωργίευα και τον κύριο Κατάινεν. Ε, θα, αυτά λοιπόν αναβάλλονται για το απόγευμα και περνάμε στο σημείο 8 η κυρία Γκρέσλε είναι η συγγήτρια αυτού του σημαντικού ζητήματος για τον καθορισμό των κανόνων που θα πρέπει να εφαρμόζεται στο Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης. Κυρία Γκρέσλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Προϋπολογισ... Κανόνες του προϋπολογισμού. Εξασφαλίζουμε τώρα την ε, εξέταση των τροπολογιών Έχουμε 76 τροπολογίες μαζί με τις δικές μου. Οι περισσότερες τροπολογίες είναι κατά κάποιο τρόπο αναδιατυπώσεις και διορθώσεις προηγουμένων τροπολογιών που είχαμε καταθέσει και όπου εμείς ως Επιτροπή είχαμε προσπαθήσει να δούμε τι είναι απαραίτητο για να προχωρήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο μέρος του πακέτου των 76 τροπολογιών. Έχουμε κάνει λοιπόν ορισμένες ε, προσθήκες για τους ε, δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αντιμετωπίσει τα θέματα της σύγκρουσης συμφερόντων με μια νέα διατύπωση, με μια νέα αιτιολογική σκέψη που καθορίζει συγκεκριμένα σενάρια για την σύγκρουση συμφερόντων και με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερος καθορισμός αυτών των περιστάσεων για να υπάρχει μια πιο μεγάλη σαφήνεια στην εφαρμογή των κανόνων αυτών. Ακολουθήσαμε αυτά τα οποία έχουν προβλέψει οι, οι διεθνείς οργανισμοί για, το, για τις περιπτώσεις που μπορεί να θεωρηθεί ένας φορέας ότι είναι μη κυβερνητικό οργανισμός διεθνούς χαρακτήρα. Ε, πάντως, δεν είχε γίνει ιδιαίτερα αποδεκτή αυτή η διατύπωση. Επίσης, έχουμε ε, προσπαθήσει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα των έμεσων ε, παραβιάσεων των δημοσιονομικών κανόνων μέσω καταπιστευμάτων και έχουμε επίσης την περίπτωση που παρουσιάστηκε στην Γκάνα όπου στην περίπτωση τριών χορηγών υπήρξε μια απάτη προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη προβλέψαμε για την περίπτωση αυτή συγκεκριμένα συγκεκριμένες ρυθμίσεις και έχουμε επίσης τροπολογίες οι οποίες αφορούν την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Θα πρέπει ο Γενικός Γραμματέας κάθε χρόνο να εκδίδει μια έκθεση δραστηριοτήτων για τα θέματα αυτά. Υπάρχει αυτή η έκθεση φυσικά στην Κομισιόν, αλλά όχι στα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούμε να γίνει και κάτι τέτοιο αντίστοιχο στα άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης έχουμε την ε, ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή Και στην έκθεση αυτή εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση του Κοινοβουλίου στην έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή μετά από συμφωνία με την Κομισιόν, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κέριο σε σχέση με την ε, διαδικασία απαλλαγή και μπορεί να γίνεται υπό το κράτος της Έχουμε επίσης και μία ε, πρόσθετη υποχρέωση για τις ε, προμήθειες οι οποίες γίνονται να τηρούν τα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα τα οποία θεωρούμε ότι ισχύουν και θέλω εδώ να εξασφαλίσω ότι γίνεται σαφές ότι η νέα οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες πρέπει να εφαρμόζεται και στα ευρωπαϊκά όργανα. Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο στα κράτη-μέλη και στους δήμους και κοινότητες και να εξαιρούνται τα ευρωπαϊκά όργανα. Επομένως πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η υποχρέωση η οποία προβλέπεται από την οδηγία για όλες τις ε, δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες. Τώρα δεν μπορούμε εμείς να λέμε όπως λένε ορισμένοι ότι αυτό δεν αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν την κατάθεση πολλών τροπολογιών για τις ε, δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες και εάν δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τότε θα υπάρξει μεγάλη οργή από τον εξωκόσμο. Η ανάγκη παραδείγματος χάρη να γίνονται διαπραγματεύσεις για την, ε, <clears throat> μετά από την ε, κατακύρωση μιας συμφωνίας και να μπορεί να γίνεται μια τροποποίηση ε, μέχρι 50% αυτών των συμβάσεων χωρίς αλλαγή της διαδικασίας, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προάγει την ε, διαφάνεια. Επομένως, εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εδραιώσουμε σωστά αυτό τον ακρογωνιαίο πυλώνα της, Ευρω της ε, ενίας αγοράς που είναι οι δημόσιες συμβάσεις και οι δημόσιες προμήθειες και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε τις απαραίτητες δεσμεύσεις οι οποίες ισχύουν για τα ευρωπαϊκά όργανα και όχι να έχουμε δημοσιονομικούς κανονισμούς οι οποίοι αφορούν μόνο τα ευρωπαϊκά όργανα. Επίσης έχουμε συζητήσει και για την τράπεζα δεδομένων που μπορεί να γράφονται σε μία μαύρη λίστα οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ε, διαπιστωθεί για τις οποίες έχουν διαπιστωθεί απάτες έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα το θέμα είναι, υπάρχουν ακόμα συζητήσεις για το αν αυτό θα μπορέσει να είναι λυσιτελές και θα μπορέσουν να λειτουργούν σωστά αυτά τα στοιχεία και σε τι θα μπορέσουν να μας ε, οδηγήσουν, γιατί πολλές φορές υπάρχει μονάχα μία μονάχα εγγραφή σε αυτή την τράπεζα δεδομένου για μία συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, Έχουμε μια πρόταση ότι θα υπάρξει ένα πάνελ, μια ομάδα εμπειρογνωμών που θα αποφασίζει ποιε εταιρείε πρέπει να εγγράφονται σε αυτή την τράπεζα δεδομένων. Και επίσης υπάρχει και η πρόταση της ε, από ΜΚΟ <clears throat> που ζητά να υπάρχει ένας μόνιμος ε, αρμόδιος για τα θέματα αυτά που να καταγραφεί και τις περιπτώσεις που υπήρξαν πρόστιμα που επευλήθηκαν. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ε, διαμοιρασμένη διαχείριση πόρων που συμμετέχει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, θα <clears throat> πρέπει να καταλάβουμε τι θα γίνει με την τροποποίηση των χρηματοδοτικών μέτρων και όλα τα κράτη-μέλη. Είναι απαραίτητο λοιπόν και για τα θέματα αυτά να υπάρχει μια έκθεση σε αιτήσιο επίπεδο. Υπάρχουν επίσης ορισμένες τροπολογίες <clears throat> για την αιτήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και, το, και για το ερώτημα τι γίνεται με την προηγούμενη ε, διαβούλευση μεταξύ του ελεκτικού συνεδρίου και του ελεγχόμενου φορέα. Και επίσης χθε προσπάθησα για τελευταία φορά να αντιμετωπίσω το ερώτημα ποια χρονικά πλαίσια θα πρέπει να, καλύπτει, να καλύπτουν οι ειδικέ εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Η συμφώνησα και με, βρήκαμε μια συμφωνία και με την Κομισιόν και θα πρέπει να γίνονται μέσα σε, 14, σε ένα διάστημα 14 μηνών και η Κομισιόν να έχει την υποχρέωση να δώσει μια απάντηση στα θέματα αυτά που αναφέρονται μέσα σε πέντε εβδομάδες. Δεν μπορεί λοιπόν να περιμένει κανείς στην Κομισιόν να ζητήσει τη γνώμη όλου του κόσμου προτού απαντήσει στα στις υποδείξεις του ελεκτικού συνεδρίου. Επίσης, για την διαδικασία απαλλαγής έχουμε ξανακαταθέσει 12 τροπολογίες οι οποίες δεν είχαν ευδοκιμήσει και αυτό αφορά την απαλλαγή για όλα τα θεσμικά όργανα και επομένως θα διασκεδάσουμε πολύ στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Έχω δει λοιπόν πέραν των δικών μου τροπολογιών και τις τροπολογίες των συναδέλφων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο. Εγώ μπορώ να έρθω σε επαφή με όλους τους συναδέλφους και να τους εξηγήσω αν βλέπω προβλήματα με τις τροπολογίες τους. Αλλά γενικά νομίζω ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση για μας. Οι κανόνες του προϋπολογισμού είναι πάρα πολύ σημαντικοί γιατί το ίμιση των υπαλλήλων της Κομισιόν εργάζεται υπό το κράτος αυτού του δημοσιονομικού κανονισμού. Πρέπει λοιπόν να περιστήλουμε την εφευρετικότητά μας και τη δημιουργικότητά μας για αυτούς τους κανόνες, γιατί είναι κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν και να εφαρμοστούν με έναν τρόπο αποτελεσματικό, γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπορούμε να έχουμε τους κανόνες όσο το δυνατόν σαφέστερους, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα ερμηνείας όπως αυτά που γνωρίζουμε ήδη με τα νομοθετικά κείμενα του παρελθόντος. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, κύριε Πρόεδρε. Ίσως θα χρειαστεί να κάνω κάποιες προφορικές τροποποιήσεις σε ορισμένες τροπολογίες, γιατί με τη συζήτηση που κάνουμε και με την Κομισιόν και με την δίκηση επίσης του Κοινοβουλίου προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι χρήσιμο και για τις διοικητικές υπηρεσίες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και προσδοκώ την περαιτέρω συζήτηση και ο κύριος ε, Γκάιερ έχει κάνει μια πολύ ωραία τροπολογία. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να περάσει και στον τριγωνικό διάλογο αφορά τον ΟΧΙΜ, δηλαδή τον Οργανισμό Σημάτων στο Αλικάντε. Και προσπαθήσαμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο ζήτησε ο κύριος Γκάιερ. Θα ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό για όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο αυτό το τομέα. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε. Επομένως, κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου και από εκεί και πέρα θα, έχουμε, θα ψηφίσουμε και θα υπάρξει και ένας ανεπίσημος ε, τριμερής διάλογος ώστε να δούμε ε, και την άποψη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος ε, Παραντή από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών που είναι διευθυντής ε, της Κεντρικής ε, Οικονομικής Υπηρεσίας έχει κάποια παρατήρηση. Πολύ γρήγορα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θεωρώ ότι ε, το προηγούμενο έργο που έχει γίνει και με την ησυχητρία την κυρία Γκρέσλε αντικατοπτρίζεται στις τροπολογίες που λάβαμε χθε το βράδυ και νομίζω ότι πολλές εξ αυτών είναι απόλυτα αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι η παρατήρηση της κυρίας Γκρέσλε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα μπορούν να το εφαρμόσουν ε, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντικό και επομένως ε, θεωρώ ότι οι τροπολογίες οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να επισημάνω τη εξή τροπολογία. Αναφέρθηκε και για το Αλικάντε. Υπάρχει ένα πρόβλημα ε, με το θέμα αυτό για τις ε, ε, υπηρεσίες και τους οργανισμούς που είναι του ΔΟΜΗ, αλλά συμφωνούμε να υπάρχει ξεχωριστός για τις, προπολογισμό για τις πράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Χαίρομαι για τις επαφές που είχε η κυρία Γκρέσλε με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή μας και είχαμε ε, ένα αποτέλεσμα, δηλαδή να γίνει δημοσίευση ε, κατά τρόπον ώστε να είναι και εύκολα να εφαρμοστεί από εμά. Να έχουμε πέντε εβδομάδε για να τη δράσουμε στη συνέχεια και να απαντήσουμε και να μπορέσουμε ίσως να απαντήσουμε από αυτού και να συμφωνήσουμε. Και όσον αφορά τη διαβίβαση τη έκθεση του ιστορικού ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, έγιναν κάποιες επαφές ε, μεταξύ μα και για αυτό το ζήτημα και θεωρώ ότι η έκθεση του ε, εσωτερικού ελεγκτού που συνήθως βέβαια είναι μόνο για το Σώμα των Επιτρόπων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να διαβιβαστεί όπως γίνεται και τώρα στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής. Κατά τα λοιπά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες τις οποίες θα εξετάσουμε από τώρα μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου με την ε, εισηγήτρια και βέβαια και στα πλαίσια των τρομερών διαλόγων που θα πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο, φαντάζομαι, προς τα τέλη Απριλίου. Ευχαριστώ. ο κύριος ε, Βεγκασκόντε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση και θεωρώ ότι όλοι θέλουμε να έχουμε κατάλληλη ρύθμιση και να υπάρχει σίγουρα διαφάνεια στις πληροφορίες. Και το αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις ευρωπαϊκές συμβάσεις. Όσον αφορά τις τροπολογίες ε, που υπευλήθησαν, υπάρχει η τροπολογία 60 και εδώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι αντικειμενικά. Δεν θα πρέπει να είμαστε υποκειμενικοί. Αποκλείονται οι προμηθευτές από μικρότερες αγορές, αλλά δεν είναι σαφές ε, τι ακριβώς εννοούμε εδώ. Νομίζω ότι από πλευρά επιχειρήσεων μπορούν να έχουμε ανεπιθύματα αποτελέσματα και να μην αυξηθεί η διαφάνεια με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Υπάρχει και το θέμα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Αυτό είναι σαφέ, μεν, αλλά θα πρέπει να είναι σαφέ και τι ακριβώς εννοούμε. Διότι μπορεί να αφήσουμε μεγάλο περιθώριο παρερμηνιών και φυσικά μπορούμε να έχουμε και ανεπιθύμητα αποτελέσματα, να υπάρχει ανεπιθύμητη πρόσβαση σε ευρωπαϊκές συμβάσεις. Δεν θέλουμε να υπάρχουν παρερμηνίες από τις ε, αρχές ε, που κάνουν τη συμβάση στα κράτη-μέλη και εμείς ως σοσιαλδημοκράτες υποστηρίζουμε το γεγονός ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι αυξημένος και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για όλες αυτές τις πληροφορίες και τις εκθέσεις ελέγχου. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια από αυτού. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανείς το λόγο. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Για την τροπολογία 60 έχω συζητήσει με πολλοί κόσμο. Γιατί θέλουμε, όπως και στο παρελθόν, να αντιμετωπίσουμε να λάβουμε υπόψη και αυτό το οποίο ζήτησε το ελεκτικό συνέδριο. Έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με εσάς. Το πρόβλημά μας είναι ακριβώς είναι η τροποποίηση στην οδηγία για τις συμβάσεις και τις προμήθειες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο αναφέρεται θα πρέπει να υλοποιηθεί γιατί εμείς πρέπει να έχουμε την απαραίτητη διαφάνεια. Και το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να κάνω είναι να παρακολουθήσω και να ενσωματώσω αυτά τα οποία έχουν γίνει σε άλλους φορείς, σε άλλες επιτροπείς. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να διοικοδομήσουμε ουσιαστικούς ε, για την ενιαία αγορά, όπως είναι η ανοιχτή πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες διαδικασίες διαγωνισμού, αυτό δεν μπορούμε να το υπονομεύουμε με το να δίνουμε απλώς μια σύμβαση με απλοποιημένες διαδικασίες στη διπλανή εταιρεία. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτό το οποίο λέτε Πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν την ισχύ των νομικών κανόνων. Οτιδήποτε κάνουμε το οποίο ε, θα έχει αποτελέσματα και για τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου γιατί υπάρχουν τώρα και νέα πράγματα τα οποία επιτρέπονται τα οποία στο παρελθόν δεν επιτρεπόταν. Αυτές οι αλλαγές λοιπόν θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή γιατί μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ανοιχτό πνεύμα και η διαφάνεια και δεν πρέπει να χαθούν αυτά. Νομίζω λοιπόν τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να ελέγξουμε προσεκτικά τι ακριβώς θα επέλθει με την τροποποίηση αυτή της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις και την προμήθεια. Αυτή τη στιγμή, τις προμήθειες αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το ξέρουμε όλο. Σας ζητώ λοιπόν να ε, Έχει την υπόψη σας ότι είμαι έτοιμη και μέσω των συνεργατών μας επίσης μπορούμε να διευκρινίσουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις ε, τροπολογίες γιατί το έγγραφο αυτό για το δημοσιονομικό κανονισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, νομίζω να το αφήσουμε το ζήτημα αυτό για σήμερα και ίσως εσείς με προφορική τροπολογία να μπορέσετε να κάνετε κάποιες ε, περαιτέρω διευκρινήσεις για να καλύψετε και τον κύριο Ιωνέσκου. Θα σας ευχαριστούμε κύριε Ισηγήτρια. Θα περάσουμε τώρα στο σχέδιο έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι επί της ουσίας είναι αρμόδια η ΕΚΟΝ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε δύο εκθέσεις ε, την Ιαρινή και τη Φθινοπορεινή και συνάδελφοι, οι συντονιστές είχαν αποφασίσει να μου αναθέσουν αυτή την έκθεση. Συνέταξα λοιπόν μια συντομότατη ομολογουμένου έκθεση όπου τονίζω πόσο σημαντικό είναι οι δημόσιοι λογαριασμοί να υπακούν στην ε, δημόσια επιταγή της ειλικρίνειας της εντιμότητας. Στη συνέχεια, χρειάζεται μια εναρμόνιση των μακροοικονομικών σενάριων επί τον οποίο εδράζονται οι προϋπολογισμοί. Στη συνέχεια αναφέρομαι στις διακοιμάνσεις που παρατηρούνται από κράτος σε κράτος και από αυτό θα έλεγα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να πλαισιώσει καλύτερα τις μακροοικονομικές τα μακροοικονομικά ερίσματα που χρησιμοποιούν τα κράτη για να καταρτήσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Στη συνέχεια, ως προς τη συμβολή των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζουμε όλοι πως υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης από πλευράς των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ποιο κομμάτι του ελλείμματος στρίκτος ε, σένσου μπορεί να αποδοθεί στις επενδύσεις ε, και αφετέρου να συνειδητοποιήσουμε μήπως υπάρχει κάποιο λειτουργικού χαρακτήρα έλλειμμα ως προς δηλαδή την εφαρμογή του προϋπολογισμού για λειτουργικά έξοδα. Είδαμε επίσης ε, με την κρίση δημοσίου χρέους ότι υπήρξαν μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ε, που δεν ελέγχονται καθόλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έπρεπε τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχουν ενεργότερα στην στον έλεγχο αυτών των χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και μην ξεχνάμε το άρθρο 13 της Συνθήκης ε, για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, χάρη στο οποίο μπορούμε πλέον ε, με θεσμοθετημένο τρόπο να εδραιώσουμε την επαφή ανάμεσα στους ευρωβουλευτές και τους εθνικούς βουλευτές και έχουμε την πρώτη ευκαιρία γι' αυτό στις 3 και 4 Φεβρουαρίου στη Διακοινοβουλευτική Εβδομάδα. Κατόπιν, Έχουμε το θέμα των μέσων που τίθεται στη διάθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και Αφεντέρου των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει. Ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα το οποίο οδηγεί σε συσσόρευση απλήρωτων λογαριασμών στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητώ ενδιάμεση αναθεώρηση δε και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου με απότερο στόχο τη μεταρρύθμιση του, πιστεύω ότι θα ήταν προσφορότερο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να συμπίπτει με την κοινοβουλευτική θητεία. Όσοι εξελέγησαν τον Μάιο λειτουργούν ε, μέσα σε ένα ε, δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο αποφασίστηκε το 2013 πρωτού διεξαχθούν δηλαδή οι τελευταίε εκλογέ του Κοινοβουλίου και ε, καλούνται να λειτουργήσουν βάσει αυτού. Ζητώ λοιπόν ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετού και έχω την εντύπωση πω τα μέλη τη επιτροπή ε, προπολογισμών θα έπρεπε ε, να προσδώσουν ιδιαίτερη σημασία στην απέτηση ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας όπως ε, επεσήμανε και το ελεγκτικό συνέδριο. Δηλαδή, πέρα από τις δαπάνες θα πρέπει να ελέγχουμε και την αποτελεσματικότητα, τις αποδόσεις. Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να κάνουν προβλέψεις ως προ τον προϋπολογισμό που θα πηχούν την πραγματικότητα και θα συνάδουν με τους στόχους που έχουν θέσει νωρίτερα Τονίζω πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα των υπολείπων προς εκαθάριση θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφέστεροι εφ' εξής. Λυπούμε διότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η συμβολή του στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνάρτηση των προσπαθειών που κάνουν για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Μα είναι εξαιρετικά ε, βολικό για τα κράτη-μέλη να ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να ε, χειριστούν καλύτερα τον εθνικό προπολογισμό και στη συνέχεια να απορρίπτουν ε, την προαποφασισμένη συμβολή του στον και λεφτή πρόταση από πλευρά μου λοιπόν. Από το έλλειμμα του εθνικού προϋπολογισμού, ας πούμε ότι έχουμε 25 εκατομμύρια απλήρωτων λογαριασμών, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάνει την εκτίμηση του ελλείμματος, του εθνικού ελλείμματος και κατά την αποτίμηση της συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Αναπτύξη να προσθέσει ένα τμήμα των απλήρωτων λογαριασμών στο έλλειμμα, το εθνικό έλλειμμα. Ε, ξέρω ότι προκαλώ με αυτή την πρόταση που κάνω, όμως για μας είναι ένας τρόπος για να επιμείνουμε για την εκαθάριση αυτών των απλήρωτων λογαριασμών. Για να είμαι λίγο αισιόδοξο και θετικός σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο Juncker, θα προσέθετα δε πως οφείλουμε να επαγρυπνούμε ως προς ε, την δημοσιονομική ε, μετάφραση των στόχων που έχουμε θέσει. Λοιπόν, πρέπει να φροντίσουμε για τα ταμεία να υπάρξει σύμπτωση των στόχων και των μέσων που αποφασίζουμε για τον προπολογισμό. Αυτές είναι οι προτάσεις, ε, συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτω μέσα στο σχέδιο έκθεσής μου, ακατόπιν έκανα και μία άλλη παρατήρηση, επί τη ουσία εννοώ πώς. Κατά τη γνώμη μου, τα κράτη-μέλη που ε, κάνουν μια επιπρόσθετη εθνική προσπάθεια σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο Juncker, τότε θα πρέπει οι κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς ε, το υπερβολικό ε, έλλειμμα να είναι πιο επίοικης. Δηλαδή, εάν οφείλεται το υπερβολικό έλλειμμα στην εξαιρετική συνδρομή ε, κάποιου κράτους μέλους στο επενδυτικό σχέδιο Juncker, να μην τιμωρείται το κράτος μέλος στη συνέχεια εδώ Μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το σχέδιο. Θυμίζω πως στις 5 Φεβρουαρίου θα ε, κληθούμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες και η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα ψηφίσει στις 23 Φεβρουαρίου τη δική της έκθεση. Ποιος θέλει να μιλήσει. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα υποστηρίζω απόλυτα. Ακόμα και τι ε, προκλητικές πλευρέ τη ε, παρουσίασή σα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτού του λογαριασμού οι οποίοι έχουν μείνει απλήρωτοι. Και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη να έχει μια προστιθέμενη αξία ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απαραίτητη αυτή ευκαμψία την οποία αναφέρατε. Χρειαζόμαστε λοιπόν να βρούμε ένα σωστό σύστημα και εδώ θα ήθελα να θέσω κάποιες δικές μου ιδέες. Γνωρίζουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτή η ολοκλήρωση απαιτεί και τα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού. Για μας δεν φαίνεται ικανοποιητικό η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να αποτελέσει θύμα του προβλήματος των εθνικών ελλημάτων προϋπολογισμού. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό θέτει ένα αμφιβόλο την φιλοδοξία που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Ο προπολογισμό μα θα πρέπει να είναι ένα προπολογισμό ο οποίο δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να πραγματοποιήσει τι φιλοδοξίε τη. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η φορολόγηση των πολιτών και θα πρέπει να αυξηθεί και το άχθο των εθνικών προπολογισμών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει και μια τροποποίηση των ιδιών πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να καταλήξουμε σε μια νέα αρχιτεκτονική η οποία θα φέρει την ευρωπαϊκή πολιτική κοντύτερα, στους πολίτες και τους ψηφοφόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πράξει τα απαραίτητα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η γνωμοδότηση θα πρέπει να είναι ένα έναυσμα για τη συζήτηση σε σχέση με τους νέους ίδιους πόρους και την υποστηρίζω ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέγει ο πρόεδρος. Ο κύριος Κολμέλ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τις ε, εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και για την ε, δέσμευση την οποία καταδεικνύεται με αυτά που είπατε. Είπατε πολλά σωστά, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε ορισμένα σημεία ήταν κάπως αντιφατικά αυτά τα οποία είπατε. Ο τίτλος της έκθεσής σας είναι «Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, δημοσιονομικών πολιτικών. Εμείς πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε αυτό υπό την οπτική γωνία του ευρωπαϊκού προπολογισμού και των εθνικών προπολογισμών. Λέτε πολύ σωστά ότι αυτοί οι προπολογισμοί πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι. Αν πρέπει όμως να γίνει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να ρωτήσω γιατί υπάρχουν τόσες πολλές τάσεις να υπονομευτεί αυτή η αρχή των ε, ισοσκελισμένων προπολογισμών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σκιώδεις προϋπολογισμοί σε πολλά κράτη-μέλη, λιγότερο ή περισσότερο. Υπάρχει η τάση επίσης οι κρατικές επενδύσεις να μην καταλογίζονται στο χρέος το κρατικό ή στο έλλειμμα. Υπάρχουν πολλά έμεσα, ε, πολλές έμεσες μορφές χρέων, χρέων που δεν ε, αναφέρονται εκπεφασμένα, παραγωγικά χάρη ε, ελλείμματα και χρέη που έχουν να κάνουν με την περίθαλψη ή με συνταξιοδότηση κτλ. Μιλάμε πάρα πολύ λοιπόν για δημοσιονομική ε, παγίωση και εδραίωση, αλλά τα αποτελέσματα είναι συχνά. Επίσης όταν αναφερόμαστε στα θέματα της ε, ευκαμψίας, εγώ πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι όταν εμείς μιλάμε για μεγαλύτερη ευκαμψία, αυτό σε σωστή μετάφραση σημαίνει μεγαλύτερη δημιουργία χρέους. Γι' αυτό θέλω να θέσω και το γενικότερο ερώτημα. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολλά πρέπει να τα συντονίσουμε αυτό, σωστό. Ίσως όμως θα πρέπει να σκεφτούμε πόσος συντονισμός στην πολιτική προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνεται και πόσο επίπεδο συντονισμού θα πρέπει να επιφέρουμε και στην οικονομική πολιτική. Έχουμε διαφορετικά προβλήματα στα κράτη μας. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια εδώ. Δεν το αφισβητώ. Γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μας και όταν ιδιαίτερα μεγάλες αυτές τις διαφορές θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και θα πρέπει να σκεφτούμε πού θα πρέπει να αφήσουμε και περιθώριο επιλογής για τα κράτη-μέλη. <clears throat> και αυτό φυσικά αναφέρεται και στο ενιαίο νόμισμα το ευρώ, το οποίο πολλές φορές κινδυνεύει από τις μεγάλες αυτές διαφορές που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Κυρία Τωμά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας πω ότι έχετε όλοι μας την υποστήριξη για τις δημοκρατικές λύσεις που υποστήριξατε στην γνωμοδότησή σας ε, και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βεβαίως, αλλά κυρίως ε, όσον αφορά τη σύμπτωση μεταξύ της ε, θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πραγματικά αποτελούν άρνηση της δημοκρατίας. Επομένως, στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου θα ήθελα να μην χρησιμοποιούμε το όρο αναθεώρηση στα μέσα της διαδικασίας, αλλά αναθεώρηση μετά τις εκλογές, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε και αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Επιπλέον, όσον αφορά τον υπολογισμό του ελλείμματος και την πρόταση την οποία εσείς ο ίδιος αποκαλέσατε ρηξικέλευθε, ε, εγώ δεν είμαι κατά των προκλήσεων. Ορισμένες φορές ε, αξίζει τον κόπο ε, να ταρακουνήσουμε λίγο τα νερά. Όσον αφορά λοιπόν αυτές τις προτάσεις, οι οποίες ε, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα, νομίζω ότι μόλις πρόσφατα είχαμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, ε, το γνωρίζουμε βέβαια, αν και μέσως έχει ε, γίνει γνωστό, ε, αλλά και άμεσα είναι γνωστό, αυτό το διαβόητο 3% δεν ήταν κατάλληλο για την περίοδο κρίσης. Χρειαζόμαστε σίγουρα ένα περιθώριο ευελιξίας ε, εν καιρό κρίσης και ίσως αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος και ίσως θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και τα υπόλοιπα προσεκαθάριση ε, σε αυτόν τον υπολογισμό του ελλείμματος από πλευράς κρατών μελών. Ε, Απ' τη μια, ναι, μεν ε, θα μπορούσα να υποστηρίξω την πρότασή σα, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι αυτό το θέμα τη ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητα ε, μα ε, ε, οδηγεί προ την άλλη κατεύθυνση επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αναθεωρεί αυτό το δόγμα το οποίο ε, βάρνει ιδιαίτερα ε, στους ώμους μας το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ο κύριος Τάγκ ε, και το ε, εισηγητή για τις πολλές προτάσεις που έκανε στην ε, γνωμοδότησή του. Έχω την Ολλανδική εκδοχή της γνωμοδότησης και ως μέλος της Επιτροπής ΕΚΟΝ θα πρέπει να σας πω ότι όντως υπάρχει έλλειψη συντονισμού στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία ε, ε, και αυτό ε, είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη υπάρχουν και διαφορέ μεταξύ χωρών μελών και αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Εγώ θεωρώ ότι ω πολιτικοί εμεί κάνουμε λίγα. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία είναι το θέμα των επενδύσεων. Είτε πρόκειται για ιδιωτικέ είτε πρόκειται για δημόσιε επενδύσει. Και εσεί, κύριε Πρόεδρε, ω συντάκτη τη νομοδότηση, ε, κάνετε μια καλή πρόταση. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του σχεδίου Juncker, το οποίο σαφώ και είναι ευπρόσδεκτο, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συνέπειες ε, των ευρωπαϊκών μέσων για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ούτε καθεξής. Εσείς πολύ σωστά λέτε ότι είναι ευπρόσδεκτες οι επενδύσεις ε, όσον αφορά το οικονομικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ε, θα πρέπει να αναλύσουμε και τις συνέπειες των επενδύσεων και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα αν ε, δω και τις προτάσεις σας, τις οποίες θεωρώ καλές, ε, μου έρχεται κατά νου και το εξής. Θα πρέπει να δούμε και τους εθνικούς προϋπολογισμού. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις, τις επενδύσεις και τις συνέπειες και αν εδώ συμπεριλάβουμε και το σχέδιο Juncker θα πρέπει να δούμε και τα θετικά και τα αρνητικά και για τους εθνικούς προπολογισμού. Διότι θα μπορούσαμε να έχουμε και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση με βάση και τις δικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Κύριε Μάνκα, για τους ίδιους πόρους. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Μόντι θα έρθει στις 5 Φεβρουαρίου. Εδώ, στην Επιτροπή μας. Euh, για να μας κάνει ένα απολογισμό της κατάστασης. Ε, τροποντινά. Όταν όμως θα ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές, ουσιαστικά θα έχουμε ε, μια επιστολή και θα είμαστε ένα κοινοβούλιο που πραγματικά θα έχει αποκτήσει μια ουσία, γιατί τώρα δεν ψηφίζουμε τους, ε, τα οικονομικά. Οι, συμβούλοι, οι Υπουργοί Οικονομικών είναι αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για αυτά τα θύματα και έχουν αυτό το δύσκολο καθήκον. Ε, είναι πραγματικό λοιπόν θέμα ε, οι ίδιοι πόροι και θα πρέπει να βρούμε και κάτι διότι ε, δεν είναι διαφορετική η ίδια η φορολογική νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος, επομένως ε, μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε φορολογία για τον άνθρακα. αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι ένα καλό εισόδημα για τους ίδιους πόρους. κύριε Κόλμερ, σαφώς πρέπει να υπάρχει συντονισμός και είναι πραγματική πρόκληση ε, να έχουμε το ίδιο νόμισμα στην υπηρεσία τέτοιων οικονομιών που είναι τόσο διαφορετικές όπως για παράδειγμα η οικονομία της Γερμανίας και της Ελλάδος. Αλλά δεν θα πρέπει εδώ ε, να κλείνουμε την πόρτα και να μην δεχόμαστε και άλλες λύσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κυριαρχία εντός εγωικών, θα πρέπει να υπάρχει και μια πραγματική κυβέρνηση που θα ασχολείται με τα οικονομικά, χρηματοπιστωτικά και νομισματικά ζητήματα. Ουσιαστικά έχουμε ένα κοινό νόμισμα, μια συνειδιοκτησία αλλά από εκεί και πέρα ε, τα κράτη-μέλη ε, παραβιάζουν τους κανόνες. Γι' αυτό ακριβώς και δεν υπάρχει κατάλληλη διακυβέρνηση. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική διακυβέρνηση. Δεν είμαι της άποψης ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να μην υπολογίζονται στα δημόσια ελλείμματα. Απλώς θα πρέπει λίγο να επαγρυπνούμε για να δούμε ε, σε τι ακριβώς ανταποκρίνεται τα ελλείμματα. Δυστυχώς υπάρχουν ελλείμματα τα οποία ε, προκύπτουν επειδή τα κράτη-μέλη δανείζονται για να ε, πληρώσουν τις δαπάνες τους. Και ε, αυτό το έλλειμμα σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι 3% αν κάποια στιγμή αλλάσουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνεται υπόψη. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα αυτό του συντονισμού, και εγώ πραγματικά θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση και καλύτερο συντονισμός. Όσον αφορά την ευελιξία, το μόνο το οποίο θα μπορούσα ίσως να φανταστώ εγώ είναι, και εδώ ίσως ανταποκρινόμαστε και σε μια ανησυχία του κυρίου Τάγκ, εάν υπάρξει από πλευράς κρατών μελών κάποια συγκεκριμένη πολιτική για το σχέδιο Juncker, Ίσως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της την ιδιαίτερη φύση υποστήριξης αυτού του σχεδίου Juncker από πλευράς κρατών μελών, γιατί βιώνουμε χαλεπούς καιρούς, η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες σε θέματα ανάπτυξης και ανεργίας και επομένως οι έκτακτες συνθήκες καλούν για έκτακτα μέτρα δεν είμαι υπέρμαχος ε, της, ε, του 3%. Είναι πολύ αυθαίρετο. Το 3% τότε υπολογίστηκε γιατί τα επιτόκια ήταν στο 5% και είχαμε ε, βάλει το όριο στο 60% του ΑΕΠ και επομένως το 60% αυτό μας φτάνει στο 3% και έτσι καθορίστηκε το 3%. Είναι το 60% του 5% αλλά χρειαζόμαστε ε, δημοσιονομική ισορροπία. Και αν έχουμε δημοσιονομική ισορροπία, τότε μπορούμε να έχουμε και πλεονάσματα στον προπολογισμό. Το 3% όμως θεωρήθηκε τότε μια καλή λύση, μια καλή δημοσιονομική πρακτική. Αν είστε στο 3% καλά τα πάτε. Αν όμως έχουμε 3% κάθε χρόνο με ένα πληθωρισμό ο οποίο ε, σχεδόν έχει εκμηδενιστεί, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει πρόοδο. Κυρία Τομά, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που θα μπορούσαμε να αποτείνουμε και θα προτείνω πολύ καλή πρόταση να κάνουμε έναν απολογισμό μετά τις εκλογές για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο πέντε ετών. Ακόμα και αν το πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα δεσμευτικό και δεν μας επιτρέπει τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε στις συγκυρίες και στην πραγματικότητα. Αυτό το προπολογισμό λοιπόν, τον υπολογισμό συγγνώμη του ελλείμματος ε, δεν είναι το θέμα των κυρώσεων αλλά αν εσείς είστε ένας οίκος αξιολόγηση. Standard Poor, Fitch κλπ. Όταν θα κάνετε αξιολόγηση τη κατάσταση μια χώρα, θα πρέπει να δείτε και ποια είναι τα υπόλοιπα τη προσεκαθάριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό εννοώ. Και η πρόκληση, αυτό το οποίο προτείνω, ε, ε, μακάρι να μπορούσατε να το προσυπογράψετε, είναι ένας τρόπος να δούμε τι έχουμε ζώσει. Στο τέλος του 2014 για να προσπαθήσουμε να πείσουμε το Συμβούλιο να μην ε, ε, βάλει στην τσέπη του τα όσα έχουν ε, περισσέψει, αλλά να αρχίσει να ε, καταβάλει τα ποσά αυτά για τα υπόλοιπα που καθάρισε. Κύριε Τάνκα, όσον αφορά το συντονισμό, συμφωνώ τους μαζί σας και για τις συνέπειες από εκεί και πέρα ε, δεν ξέρω αν τα κράτη-μέλη λαμβάνουν υπόψη και το θέμα αυτό στον προπολογισμό τους, αλλά λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ίσως να προσθέσει στο έλλειμμα που υπολογίζει και το δικό του το μερίδιο για τα υπόλοιπα αυτά που σε Ο κύριος Δονατό, οι προτάσεις σας... Ε, ε, είναι όλες ε, τιμωρητικές. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο δέλεαρ ώστε ε, να μπορέσουν να προσπαθήσουν τα κράτη-μέλη να μειώσουν τα ελλείμματα. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ευαλιξία για να είναι λίγο ισορροπημένα τα πράγματα. Ο Πρόεδρος. Αν έχετε εσεί τροπολογία το, η οποία θα αποτελέσει δέλεαρ, είμαι διατεθειμένο να τη δεχτώ. Αλλά τα ίδια τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη για να έχουν μια κοινή νομισματική κυριαρχία. Θεωρώ λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φύγουν από αυτή την ευκολία του window dressing αν θέλετε. Δηλαδή ε, να υπάρχει ε, μια σαφής εικόνα, μια ειλικρίνεια στα δημόσια οικονομικά. Και όταν ξέρουμε την αλήθεια τότε θα μπορούμε να λάβουμε σωστές αποφάσεις και τελικά ε, ε πολλές φορές ε, αναγκαζόμαστε ε, να βρεθούμε ενώπιον της κατάστασης και να δεχτούμε ότι είναι ζωφερή. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να αρνούμαστε την πραγματικότητα και να δεχτούμε την πραγματικότητα. Ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως θα μπορούσαμε να το θέσουμε σε γραπτή μορφή αυτό και να υπάρχει ε, και κάποια σαφέστερη διαδικασία για τη μαύρη λίστα. Για τους ίδιους πόρους δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη από μόνα τους δεν μπορούν να αποφασίσουν για τους ίδιους πόρους. Αυτό είναι μια υπόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με για τα θέματα των δύο πόρων και να τονίσουμε ότι δεν έχει κλείσει η συζήτηση, αλλά είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε περισσότερο. Θα εργαστούμε για το θέμα αυτό. Στις 5 Φεβρουαρίου καταρχήν. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα ερχόμαστε στις ψηφοφορίες. Και πάμε στο σημείο 14 καταρχήν, στην έκθεση του σημείου 14. Είναι η ετήσια έκθεση του, της υπάτης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξωτερικά θέματα, την πολιτική ασφάλειας. Η συγητής είναι ο κύριος Τάραμβ. Υπάρχει εδώ η τροπολογία υπαριθμών 1. Ο εισηγητή είναι υπέρ αυτή τη τροπολογία. Ποιοι υποστηρίζουν αυτή την τροπολογία επίση. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Μάλλον ποιο είναι κατά. πούμε, Δεν υπάρχει κανεί κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 7 υπάρχει η τροπολογία υπαριθμών 2 με ψήφο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ο κύριος Ταραντ είναι υπέρ, ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος. Ευχαριστώ. Κατά. Μία, μία ψήφος κατά. Αποχές. Μάλιστα. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας. Επίσης το υποστηρίζει ο κ. Σταράν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Τρεις ψήφι κατά. Τέσσερις κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα υπέρ ο κύριος Στάραντ. ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Σας ζητήσω να ε, κάνετε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεν λειτουργήσε. Ξαναρχίσουμε. Εντάξει. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Παράγραφο 8. Η τροπολογία υπαριθμών 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα το υποστηρίζει ο εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, πάλι το υποστηρίζει ο εισηγητής, ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα, παράγραφος 9, τροπολογία 4, δεν το υποστηρίζει ο συγητής, ψηφί υπέρ. Μα θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 22-7 και τρεις αποχές. Το σύνολο του κειμένου πως έχει τροποποιηθεί Ποιος θέλει να λάβει το λόγο, κύριο Σαλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω μόνο να σας πω πως ο κύριος Ντεπρέ, που είναι συγκεκριτής για τα υπόλοιπα τμήματα, δεν έχει ενημερωθεί για αυτές τις τροπολογίες. Και νομίζω ότι εκφράζω την άποψή του και τη δικιά μου σίγουρα όταν λέω πως ζητήματα που σχετίζονται με το 2016 για το 2016 ε, θα πρέπει να είναι γνωστά στον εισηγητή για το 2013. να μπερδεύουμε λίγο τα δύο ζητήματα εδώ. Euh, Έχει γίνει η ψηφοφορία όμως. Ε, ναι, αλλά θέλω να το έχετε ε, υπόψη σας, ε, διότι έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Κάποια σχετίζονται με το 2016 και δεν μπορούμε να τα μπερδεύουμε με αυτή την έκθεση που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό του 2013. Πρόεδρος, λαμβάνουμε γνώση της δήλωσής σας, όμως έχει γίνει ψηφοφορία και ζητώ από την Επιτροπή να ψηφίσει για το σύνολο με ονομαστική ψήφο. Έχουμε πρόβλημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίθηκε με 27 ψήφους, 2 ε, και 3 αποχές. Σε πόλη τώρα. Τι γίνεται με την ε, ε, προσέγγιση της ΕΠΟΛ και Europol, ξέρετε, κύριε Γκάιερ, stand by. Τροπολογία 3 είναι υπέρ ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε με 18 προς 3. Τροπολογία 4 για το άρθρο 24 είναι υπέρ ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Και για τα παραρτήματα και τα εκτιμώντας 12-1 ε, είναι παρουσιογητής υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Αιτιολογική 15 τροπολογία 2 είναι υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Πρέπει να διαβάσετε την προφορική τροπολογία. Κατέπεσε. Ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη γενικότερη ανάλυση της διοικητικής συνεργασίας ανάμεσα στους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τους τομείς όπου θα μπορούσαν μελλοντικά να υπάρξουν τέτοιες συνεργασίες. Κύριε Γκάιερ, είστε υπέρ, ποιοι είναι υπέρ αυτής της προφορικής τροπολογίας. Ευχαριστώ κατά. Αποχές δεν υπάρχουν. Το σύνολο τώρα, παρακαλώ, υπέρ. Α, ναι, πρέπει να γίνει ηλεκτρονική, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Μου σφυρίζουν εδώ ότι υπάρχει ένας υπεράριθμος του ΕΛΚ. Ωραία. Λοιπόν, 17 ψήφοι προς 13 και 4 αποχές. Εγκρίθηκε το κείμενο. Περνάμε τώρα στο ε, σχέδιο του κυρίου Ταχά. Πρόκειται για την απόφαση του Συμβουλίου και τη σύναψη μιας ε, συμφωνίας ε, ε, εταιρικής σχέσης για την Αλία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την δημοκρατία της Σενεγάλης. Δεν έχουμε τροπολογίες, επομένως ποιο ψηφίζει υπέρ του κειμένου. Α, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Non, c'était pas forcément l'appel nominal, mais ça fait rien. Le vote est clos. Πέρασε η ψηφοφορία. Un vote sur ah Α, πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε τη συμφωνία ε, ε, εταιρικής σχέσης. Ποιοι είναι υπέρ της συμφωνίας. Είναι ε, υπέρ ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Μπορείτε να κατεβάσετε τα χέρια σας. Ποιος είναι κατά. Δεν υπάρχουν ούτε αποχές, επομένως εγκρίνεται. Και τώρα ε, τη γνωμοδότηση του κυρίου Ταρά. Εδώ ε, ηλεκτρονικά. est Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε est ψηφοφορία. 33 ε, ψηφίσαντες, 33 υπέρ. Εξαιρετικά. Τώρα, περνάμε στο σημείο 17. έκθεση του κυρίου Ντεπρέ για την ε, μεταφορά πιστώσεων, κάποια θέματα που βρίσκονται σε κάποιους τίτλους στο τέλος του 2014 και ε, μας έχει ζητηθεί γνωμοδότηση ώστε να μπορέσουν να ε, καλυφθούν κάποια υπόλοιπα προς και να μειώσουμε το υπερβολικό έλλειμμα που γνωρίζετε. Έχετε το κείμενο. Ο κύριος Αλή που εκπροσωπεί το κύριο Ντεπρέ έχει κάτι να μας πει. Όχι. Έχετε το κείμενο. Η μείωση αυτή αφορά 36 γραμμές προπολογισμού, 36 τίτλους. Έχουμε 5 τίτλους ενισχύονται κάποιες από τις εκκρεμότητες, 3 ε, γραμμές προπολογισμού εδώ, 9 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη του Ευρωπαϊκού Ελευτικού Ταμείου, 466 ε, για το Ταμείο Συνοχής εκατομμύρια και 4,6 εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Επιστροφής Προσφύγων και Επαναπατρισμού. Και θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι βάσει και των όσων έχουμε υποστηρίξει ως συγκεκριμένη γραμμή προπολογισμού, η επιστροφή των ποσών αυτών στο Ταμείο Συνοχής ε, είναι καλό νέο κατά την άποψή μας. Ευχαριστώ. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν αυτής ε, της πρότασης. Τα ευχαριστώ. Κατά. Δεν βλέπω κανένα κατά. Δεν υπάρχουν ε, ούτε αποχές. Επομένως υπερψηφίζονται αυτές οι μεταφορές κονδυλίων. Σημείο 19. Άλλα τμήματα. Η κυρία Χόλμα η ερνησυγήτρια. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο εδώ. Και με αυτό ολοκληρώνουμε. Και ολοκληρώνουμε και γέρος. Θα διακόψουμε λοιπόν τώρα τις εργασίες μας και θα συνεχίσουμε στις 3 σήμερα το απόγευμα με την ακρόαση του κυρίου Κατάινεν και της κυρίας ε, Γεωργίεβα για το σχέδιο Juncker και για το σημείο 1 που επιτρέπει ε, την εφαρμογή από τον Ιούνιο του πρώτου τμήματος του σχεδίου 2 και θα παρουσιάσει και το ε, δεύτερο τμήμα η κυρία Γεωργίευα. Στις 3 η ώρα λοιπόν και μετά τη συνεδρία της Επιτροπής θα συνεδριάσουν οι συντονιστές.